Ε, και τα εγκεκριμένα κείμενα υπάρχουν ε, και θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν παρατηρήσεις σε σχέση με τα χθεσινά πρακτικά. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο.